Έχουν ε, το όνομα Χωριάν Πεστέιρο που ήταν ε, καθηγητής ε, δεοντολογίας, ηθικής και ήταν ένας καθηγητής ο οποίος πέθανε στις φυλακές του Φράγκο από συψεμία. Να δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφό μας Εμέρ Κοστέλου. Ευχαριστώ.